Buonasera. Καλησπέρα. Η συνεδρίασή μας ε, θα πρέπει να γίνει με την ύψιστη σοβαρότητα, δεδομένου ότι είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Έχουμε απαρτία και αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν είναι παρόντες λόγω της προεκλογικής εκστρατείας. Εξάλλου, τα ζητήματα που έχουμε συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη δεν είναι τόσο σημαντικά όσον αφορά την οικοδόμηση της Ευρώπης. Να σας ενημερώσω ότι έλαβε χώρα η συνεδρίαση των συντονιστών. Εδώ θα το εξετάσουμε αυτό πρώτο αντί για τελευταίο για να σας δώσω κάποιες πληροφορίες που θα καθορίσουν την ημερήσια διάταξη. Συνιστούν οι συντονιστές στην Επιτροπή να περιοριστούν σε ερμηνεία των άρθρων 165 και 159 του κανονισμού βάσει επιστολής του υπογεγραμμένου που έχουν λάβει του επιφανόμενου που έχουν λάβει όλοι οι παρόντες. Αυτό είναι το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Επίση η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν έπρεπε να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη τα αιτήματα ψηφίσματος των συναδέλφων Κλάς και Μαριλεπέν για έναν πολύ απλό λόγο. Ζητούν την κατάργηση θεσμικών οργάνων, πολύ απλά, που ε, αποτελούν αντικείμενο των συνθήκων. Συνεπώς εμεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αυτή τη στιγμή. Για τον ίδιο λόγο ουσιαστικά οι συντονιστές πρότειναν να μην συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη το αίτημα του συναδέλφου Μάρτιν να παρουσιάσει ένα έγγραφο εργασίας για το ζήτημα της απόσχησης ενός κομματιού μιας χώρας. Δεν μας έχει υποβάλει κανένα έγγραφο, δεν ξέρουμε περί τι να συζητήσουμε. Φυσικά έχει την ελευθερία να παρουσιάσει κάποιο έγγραφο εφόσον το επιθυμεί και να το δημοσιοποιήσει, αλλά δεν μπορεί να έχει την έγκριση ούτε έμεσα της Επιτροπής αυτής. Έτσι λοιπόν θεωρήθηκε ομόφωνα μεταξύ των συντονιστών ε, ότι δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να παρέμβει για τις ανακοινώσεις αυτές ο συνάδελφος κ. Μπρόγκς. Ευχαριστώ. Κατάλαβα καλά. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ εδώ πέρα κάτι το οποίο απαιτεί αλλαγή της συνθήκης. Αν θυμάμαι καλά, ε, ο κύριος ε, Ρανκέλ είχε παρουσιάσει μια έκθεση στην οποία πρότεινε ένα προεδρικό σύστημα ε, και όχι ένα πρωθυπουργικό ας πούμε και το είχαμε συζητήσει οπότε δεν ήξερα ότι είναι κατά του κανονισμού το να συζητάμε πράγματα που απαιτούν αλλαγή της συνθήκης αλλά αν κάνω λάθος διορθώστε με Ο κύριος Δάφ. Μπορούμε να συζητήσουμε τροποποίησεις των συνθηκών στην ε, Επιτροπή μας αυτή και στο κάτω-κάτω αυτός είναι και ο κύριος σκοπός της Επιτροπής αυτής. Είναι όμως σημαντικό να βάζουμε τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο τους. Να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή όλες τις συνταγματικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε την ομοσπονδιακή πορεία και να να μην ε, επιλέγουμε από εδώ και από εκεί διάφορα κομματάκια ανεξάρτητα από το γενικό θεσμικό οικοδόμημα. Αυτό θα ήταν εσφάλμα. Ευχαρίστως. Στα πλαίσια της συνέλευσης, η οποία έχω πιστεύω ότι θα λάβει χώρα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ευχαρίστως να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση για τον ε, λόγο ύπαρξης, τη λειτουργία, το κόστος και τις εξουσίες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. Με κάθε σεβασμό. Πιστεύω ότι δεν είναι τώρα ο κατάλληλος χρόνος, η κατάλληλη στιγμή δηλαδή, ο κατάλληλος χώρος για να κάνουμε μια τέτοια τόσο ριζοσπαστική συζήτηση. Είναι επίση σημαντικό να μεταχειριζόμαστε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάθε σεβασμό. Όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών, αν λάβουμε υπόψη μας το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φαίνεται να είναι περισσότερο πόλεις μαζί, πολύ περισσότερο από ότι μια συνομοσπονδία κρατών, τότε θα έπρεπε αντίθετα να ψάξουμε να βρούμε τρόπους για να αναβαθμίσουμε το ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών. Πάντως, όπως είπα και πριν και με κάθε σεβασμό, πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή ούτε ο κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάλλον θα συμφωνήσω με τον κύριο Νταφ. Εντάξει, αναφερθήκαμε σε αλλαγέ στη συνθήκη. Μα εδώ περισσότερο πρόκειται για τον κανονισμό, για αλλαγέ στον κανονισμό, αν πάση περιπτώσει. Αν αυτό το θέμα τεθεί, το μέλλον δηλαδή των δύο αυτών θεσμικών οργάνων, τότε θα πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας πολύ γενικότερη συζήτησης που θα αφορά τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανατομία της, τη λειτουργία της, και σίγουρα ούτε και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ο κατάλληλος χώρος ή χρόνος για να γίνει η συζήτηση αυτή. Μάλλον θα πρέπει να την κάνει η επόμενη εντολή, η επόμενη θητεία, το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι περίεργη η διαδικασία αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι ο σωστότερος τρόπος για να αρχίσει μια τέτοια συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να το αφήσουμε για το επόμενο κοινοβούλιο, για την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέπετε μια γρήγορη ερώτηση προς τον κύριο Νταφ. Στην πρώτη σας πρόταση φαίνεται πως υπονοείτε πως εντάξει να συζητήσουμε αλλαγές της συνθήκης αρκεί να οδηγούν σε ομοσπονδιακή κατεύθυνση και όχι στην αντίθετη. Τι να σα πω, μπορεί να κατάλαβα και, και λάθος είμαι, κακός. Όχι, όχι. Ε, Πλάκα σας έκανα κύριε Μπρόντς. Σας πείραζα. Σε ένα ομοσπονδιακό κατασκεύασμα οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες ε, μπορούν να ρέουν και προς τα ανάντι και προς τα κατάντι. Va bene, possiamo... Ωραία λοιπόν. Α, παρακαλώ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φίλιπ Κλάις, ένας εκ των συντακτών του ψηφιτών ψηφισμάτων και συμπτωματικά με ενημέρωσαν για το ότι είναι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Αλλά βεβαίως εγώ θα ήθελα να γίνει μια συζήτηση για τα ψηφίσματα αυτά. Αυτό δεν έχει ούτε μία σχέση με το εάν είναι κανείς ε, ευρωσκεπτικιστής ή ευρωκριτικός ή ευρωομοσπονδιακός. Λέμε να γίνει μια αξιολόγηση διαφόρων ε, υπηρεσιών, θεσμικών οργάνων και λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε όπως είπα, κάποια ψηφίσματα που υποβάλαμε εγώ και η συνάδελφος, δύο από αυτά είναι προς συζήτηση, αλλά νομίζω πως είναι προς το συμφέρον όλων, ανεξαρτήτως της ε, στάσης τους, να γίνει αυτή η συζήτηση και η αξιολόγηση για την λειτουργία αυτών των θεσμικών οργάνων και όχι μόνο για την ΟΚΕ και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αλλά μπορούν νομίζω να τεθούν ε, κάποια ερήματα, κάποια ερωτήματα. Π.χ. για την Επιτροπή των Περιφερειών φαίνεται πως έχουμε ένα μίνι ε, φωτοαντίγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι οργανωμένοι σε κοινοβουλευτικές ομάδες με γραμματείες ομάδων, ταξίδια ομάδων συνεργάτες ομάδων Νομίζουμε λοιπόν πως αυτό είναι το σωστό και τελικά ποιο αποτέλεσμα έχει η λειτουργία της ε, Επιτροπής των Περιφερειών. Εγώ πρέπει να σας πω πως προσπάθησα κάποιες φορές ε, να διαβάσω αυτές τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών που μας στέλνουν πριν τις ψηφοφορίες. Αλλά πρόκειται για φωτοτυπία των όσων αναγράφονται εδώ πέρα, ίδιες ακριβώς θέσεις από τα ίδια ακριβώς κόμματα και η προστιθέμενη αξία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Γι' αυτό θεωρώ πως πρέπει να συζητήσουμε πώς ε, λειτουργούν αυτά τα θεσμικά όργανα. Έχουν κάποια χρησιμότητα, έχουν κάποια σημασία. Ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξής τους. Είναι σημαντικά νομίζω αυτά τα ερωτήματα και είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και που να κοιτάει με μια κριτική ματιά την προσθέμενη αξία τέτοιων θεσμικών όργανων όπως η Επιτροπή των Περιφερειών. Ζήτησε το λόγο ο συνάδελφος Νταφ. Κύριε Κλέες, δεν προτείνω να μην το συζητήσουμε το μέλλον αυτών των δύο επιτροπών. Μάλιστα, η πρώτη δουλειά που έκανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 1974 μια μελέτη για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για το μελλοντικό σκοπό ύπαρξής της. Δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού τότε και υποψιάζομαι δεν θα καταφέρουμε ούτε τώρα. Αλλά η πρότασή σας κάνει έκκληση για κατάργηση αυτών των δύο επιτροπών. Κάνει πρόταση για κατάργηση και όχι για μια σκέψη και μελέτη για μια συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται Δεν νομίζω ότι η διάσκεψη των Προεδρών δεν θα συμφωνούσε με την άποψη των συντονιστών. Στην παρούσα φάση του Κοινοβουλίου δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα. Εκεί νομίζω ότι το όλο ζήτημα και εκεί θα παραμείνει μέχρι το φθινόπωρο. Yes, thank you, Chair. Just follow on με ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να συνεχίσω και την επιχειρηματολογία. Νομίζω ότι αυτό για το οποίο συζητάμε ουσιαστικά είναι έλεγχος οικονομικός ενδεχομένως αυτών των δύο επιτροπών και είναι μάλλον ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί στη συνέλευση παρά υπό αυτή την οπτική γωνία που προτείνεται εδώ και γιατί αυτούς τους δύο οργανισμούς, θεσμικού, αυτά τα δύο θεσμικά όργανα και όχι άλλα, δεν βλέπω για ποιο λόγο. Και δεύτερον, θεωρώ ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να προτείνουμε ευθύ εξ αρχή την κατάργηση ω αφιτηρία. Αντίθετα, θα πρέπει να δούμε τη λειτουργία, τη διάρθρωση, το σκοπό ύπαρξη αυτών των δύο θεσμικών οργάνων και θα, σαφώς είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί στη συνέλευση και όχι σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. I think this is a, a good opportunity for me to point out we spent the last quarter. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξέρουμε ότι εδώ συζητάμε ένα τέταρτο για ένα θέμα για το οποίο συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να βάλουμε και άλλη μια πρόκληση. Να, έχω εδώ δίπλα μου, ορίστε, τη ζητώ μάλιστα και να σηκωθεί. Είναι η Λίζ Μπάκλ. Όπως βλέπετε, η Λίζ δεν έχει χέρια ουσιαστικά, τα άνω μέλη. Η μητέρα της πήρε ένα φάρμακο κατά την εγκυμοσύνη, το Φελίντε Μάι το οποίο είναι μια γερμανική εταιρεία της Greenenthal, το φάρμακο αυτό, και δημιούργησε προβλήματα. Όλοι όσοι βρέθηκαν στην κατάσταση που βρίσκεται και λύζει σήμερα γεννήθηκαν τη δεκαετία του 50 και φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστικό αυτού του φαρμάκου. Χρειάζονται περισσότερη προσοχή, χρειάζονται και περισσότερα χρήματα εννοείται για να έχουν τη μέρη που του χρειάζεται. Η εταιρεία Greenenthal λοιπόν, εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε τη σήμερα και η γερμανική κυβέρνηση επίση, η οποία έχει και την ευθύνη. Τι, η ευθύνη δεν είναι μεγάλη. Για το Ηνωμένο Βασίλειο μιλάμε για 30 cents το χρόνο ανά γερμανό φορολογούμενο που θα μπορούσε να είναι 50 το χρόνο αν βάλουμε και όλες τις αντίστοιχες ασθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να ενημερωθεί γι' αυτό ο κόσμος και ιδίως εδώ τα μέλη της Επιτροπής μας. Ναι, για αυτή την τελευταία παρέμβαση συμφωνώ και συμμερίζομαι τα όσα είπατε, αλλά δεν υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη αυτά τα ζητήματα ως θέμα και δεν αποτελεί κομμάτι της αρμοδιότητας αυτής της Κομισιόν, Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι αποτελεί πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν μπορούν να βρουν λύση για κάτι τέτοιο, για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η σημαία πίσω σας, για ποιο λόγο. Μα νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό είναι και πρόβλημα των επιμέρους κρατών μελών. Καταρχάς και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έλεγα σκόπιμο θα ήταν να μην επιμείνετε. Σαφώς συμμερίζομαι ε, το ε, θέμα που ε, βασάνισε την κυρία και φυσικά θα πρέπει να βοηθούν τα κράτη-μέλη. Συνεχίσουμε όμως τη συζήτηση για το θέμα της πρότασης, των προτάσεων ψηφίσματος ε, για την κατάργηση. κυρία Πέτροβιτς ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους προλαλήσαντες. Να συμπληρώσω και εγώ κάποια πράγματα. Θεωρώ πως μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις εδώ πέρα για τη λειτουργία των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως επίσης και για την Επιτροπή των Περιφερειών και την ΟΚΕ. Αλλά ανεξαρτώς του αν είναι εδώ το κατάλληλο μέρος να γίνει αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε το πότε θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι σήμερα η κατάλληλη ημέρα. Νομίζω μπορούμε να αναβάλουμε τη συζήτηση για το φθινόπωρο, θα έλεγα εγώ, για αυτά τα δύο. Και να σας παραπέμψω, να επισημάνω πως έχουμε εδώ πέρα επισκέπτες από την Κροατία, νεαρούς, οι οποίοι αναμένουν την συζήτησή μας. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής θα μπερδευτούν μόνο με το πώς γίνεται η συζήτηση εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σύντομα για κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν. Δεν είναι ε, η δική μου επειδή η δική μου εφετηρία είναι πως δεν χρειάζονται αυτά τα θεσμικά όργανα ε, και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να γίνει συζήτηση. Πράγματι, εγώ είμαι αρνητικός γιατί εμφισβητώ την χρησιμότητά τους. Αλλά Βεβαίω, αν κάποιο έχει επιχειρήματα για το αντίθετο, ευχαρίστω να τα ακούσω. Αυτό είναι το, το νόημα. Αυτή είναι η πρόταση που ήθελα να κάνω. Να γίνει δηλαδή μια συζήτηση για αυτό το πράγμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι κρίμα ότι προσπαθεί να βρούμε διάφορα διαδικαστικά ε, και να συγκληθεί ολόκληρη συνέλευση για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Όχι, μια χαρά μπορούμε ως Κοινοβούλιο να συζητήσουμε τη λειτουργία των άνω θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Εγώ θα πρότεινα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Οι συντονιστές ε, πρότεινα να δεν κάνω λάθος να μην δώσουμε συνέχεια σε αυτές τις δύο προτάσεις ψηφίσματος όχι διότι αντιτίθενται επί της ουσίας. Εγώ πρώτος το επαναλαμβάνω και το είπα ήδη στις συνεδρίες των συντονιστών, θεωρώ ότι είναι σοβαρές και βάσιμες και σωστά αιτιολογημένες οι προτάσεις αυτές. Ε, μπορούμε να πούμε και ε, κάτι από τον λατινικά ότι δεν χρειάζεται να διπλασιάζουμε μέσα όταν δεν είναι απαραίτητε, αλλά σίγουρα, όπως είπα στον κύριο Νταφ, θα πρέπει να ζητηθούν σε ένα άλλο πλαίσιο το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε σήμερα. Μπορούμε να το κρατήσουμε ως επισήμανση του προβλήματος αυτού για το επόμενο κοινοβούλιο. Γιατί το κοινοβούλιο δεν μπορεί να τροποποιήσει τις συνθήκες. Ε, αναφέρεται αυτό στο άρθρο 48. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως ε, θα το συζητήσουμε όμως μετά. Εφόσον συμφωνείτε έχει προβληθεί μια θεματική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης για το επόμενο κοινοβούλιο θα αποτελέσει ουσιαστικά δότημα για το επόμενο κοινοβούλιο για το ποιο, ποια μελλοντικά ζητήματα θα συζητηθούν και μπορεί να συμπεριληφθεί εκεί διαφορετικά δεν μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε εδώ για αυτό το θέμα στην παρουσία φάση αυτή ήταν η απόφαση της πλειοψηφίας κάποιες άλλες ανακοινώσεις σημαντικές αφορούν την εργασία για τα πολιτικά κόμματα που μας απασχόλησε τόσο καιρό, όπως γνωρίζετε όλοι, όπως θα θυμάστε. Το τελικό κείμενο του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα εγκρίθηκε 18 Μαρτίου αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστική τελειοποίηση του κειμένου από τις γραμματείες του Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο. Πρόκειται για μια αναθεώρηση που χρειάζεται χρόνο και προβλέπεται η εργασία αυτή να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαμεθήμερο του Μαΐου. Τι θα συμβεί μετά, εφόσον οι τροποποιήσεις είναι επιφανειακές, τίποτα, δεν έχουμε πρόβλημα. Αν χρειάζονται τροποποιήσεις που αφορούν την ουσία, εκεί θα απαιτείται η συζήτηση να γίνει στην Επιτροπή μας, η οποία Επιτροπή μας θα πρέπει να ε, υποβάλει να καταθέσει μια έκθεση στην Ολομέλεια. Όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν αυτή τη στιγμή σε αυτήν εδώ τη θητεία προφανώ. Υποθετικά είναι τα σενάρια που σας ε, παρουσιάζω σε περίπτωση που γίνουν προτάσεις διορθώσεων επί τη ουσία και όχι μόνο επί γλωσσικών ε, θεμάτων, ουσιαστικά γλωσσικών. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ουσιοδών τροποποιήσεων θα χρειαστεί να παρέμβουμε και να το ζητήσουμε από την Ολομέλεια. Αυτό δεν θα είναι δυνατόν σε αυτή τη θητεία διότι η επόμενη Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα είναι και η τελευταία. Η πρόταση λοιπόν είναι σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με μια πρόταση τροποποίησης επί της ουσίας θα ακολουθήσουμε μια γραπτή διαδικασία ώστε το επόμενο κοινοβούλιο να μπορέσει να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό αμέσως μόλις εκλεγεί στις πρώτες του συνεδριάσεις και όχι υπερβολικά καθυστερημένα. Αυτή είναι η πρόταση που έχω να σας κάνω, δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε. Εφόσον συμφωνείτε θα το θεωρήσουμε ότι αποφασίστηκε η άλλη ανακοίνωση βασίζεται στο αίτημα του θεματικού τμήματος να λάβει άδεια, να διοργανώσει τον επόμενο Σεπτέμβριο ένα σεμινάριο για τις μελλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης που αναμένουν το επόμενο κοινοβούλιο. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στις συνταγματικές υποθέσεις πρέπει να πω ότι και άλλες επιτροπές έλαβαν το ίδιο αίτημα όπως η Επιτροπή Γιούρη και η Επιτροπή ε, ΦΕΜ και έχουν δώσει ήδη άδεια στο θεματικό τμήμα να διοργανώσει ένα σεμινάριο για το θέμα αυτό. Όχι για αυτό το θέμα, για θέματα που εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα. Μα ζητούν λοιπόν να τους δώσουμε την άδεια να προετοιμάσουν ένα σεμινάριο για τις μελλοντικέ προκλήσεις. Και εγώ θεωρώ ότι σκόπιμο θα ήταν γιατί σε τελική ανάλυση ε, σημεία όπως αυτά που εμφανίστηκαν εδώ στη συζήτηση θα μπορούσαν να αναφερθούν επί τη ευκαιρία τέτοιων σεμιναρίων. Ε, συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση είναι συζητήσεις. Ε, αν συμφωνείτε λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διαφωνία. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε την έγκρισή μα. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι την επόμενη Πέμπτη από τις 9 μέχρι τις 12.30 το πρωί θα λάβει η χώρα η δημόσια ακρόαση για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών δυνάμει του άρθρου 11 της συνθήκης της Λισαβόνας που αναφέρει τον επαρκή αριθμό ατόμων και χωρών ώστε να λάβει χώρα μια τέτοια ε, ακρόαση. Η ακρόαση λοιπόν θα καθοδηγηθεί από τις Επιτροπές ε, Νομικών Υποθέσεων, Βιομηχανίας και Έρευνας, Ανάπτυξης και φυσικά από την Επιτροπή Αναφορών. Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν κληθεί να συμμετάσχουν. Θεωρώ ότι οι βουλευτές της Επιτροπής ΑΤΚΟ πρέπει να προσκληθούν ιδιαίτερα σε αυτή την ακρόαση, αν τι άλλο, διότι σε αυτήν εδώ την Επιτροπή ε, μελετήθηκε το νέο ο νέος κανονισμός. Υπάρχουν περαιτέρω ε, τροποποιήσεις για τον κανονισμό ίδρυσής του, όχι μόνο όσον αφορά το περιεχόμενο του αιτήματο, αλλά και για τη μεθοδολογία. Καλό θα ήταν λοιπόν να βρίσκονται εκεί οι, τα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Σας ε, προσκαλώ λοιπόν να συμμετάσχετε στην ε, ακρόαση αυτή την επόμενη Πέμπτη από τις 9 μέχρι τις 12.30. Ξέχασα κάτι. Πρόκειται για μια δημόσια ακρόαση και θα έχει μεγάλη προσέλευση. Η γραμματεία λοιπόν σας παρακαλεί μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα να ενημερώσετε την γραμματεία ότι προτίθεστε να συμμετάσχετε εφόσον προτίθεστε. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων 10 και 10 Φεβρουαρίου τα πρώτα πρακτικά και 10 Μαρτίου 2014. Τα έχετε στη διάθεσή σας σύμφωνα με ναι, ό,τι ήθιστε θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Το σημείο τώρα που θα συζητήσουμε για να λάβουμε μια απόφαση αφορά την ερμηνεία του άρθρου 166 και του άρθρου 195 του κανονισμού. Λοιπόν, για να σας δώσω μια σύνοψη. Όπως γνωρίζετε, εμείς πρόσφατα εισήγαμε μια τροποποίηση στον κανονισμό. Η τελική ψηφοφορία για οποιαδήποτε έκθεση, νομοθετική ή μη, είτε στην Ολομέλεια είτε σε Επιτροπή πρέπει να γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία. Ήδη το εφαρμόζουμε. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, ε, ε, η κυρία Ρέγνερ δεν είναι εκεί, αλλά μας ζητά να εξετάσουμε κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μια γνωμοδότηση που θα επιτρέπει μια ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή μυστική ψηφοφορία, για θέματα που αφορούν άρση βουλευτική ασυλία. Βάσει του επιχειρήματο ότι σε τέτοια θέματα άρση ασυλία αποφασίζουμε για συγκεκριμένα άτομα και υπάρχει κάποια αρχή στον κανονισμό βάση τη οποία ο κατονομασία ατόμων πρέπει να γίνεται με ψηφοφορία μυστική. Τώρα, αυτή η διαδικασία απόφασης κατά πόσο θα έρουμε ή όχι την ε, ασυλία απαιτεί κάποια συζήτηση και κλεισμένο των θυρών και ψηφοφορία επίσης και κλεισμένο των θυρών. Συνεπώς αποτελεί εξαίρεση στην αρχή της δημοσιοποίησης που θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί και στα ονόματα των ανθρώπων που ψήφισαν ε, υπερικατά. Δύναμη του άρθρου 7 περί ασυλίας αναφέρεται ότι τα έγγραφα πρέπει να διατηρούνται απόρριτα και όχι να δημοσιοποιούνται. Διάφορες λοιπόν τέτοιες αναφορές μας επιτρέπουν να πούμε ότι η ψηφοφορία περί ασυλίας ε, είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται μυστικά και όχι ονομαστικά. Αυτό απαιτεί παρέμβαση της Επιτροπής μας. Προτείνω λοιπόν να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Αν συμφωνείτε θα πρέπει να εκδώσουμε μια γνωμοδότηση ερμηνευτική μέσω μιας επιστολής. Με αυτό που σας διανύμαμε και σας το διαβάζω, οι διατάξεις των άρθρων 166-167 παράγραφος 1 και 195 παράγραφος 3 για την ψηφοφορία για την ονομαστική ψηφοφορία δεν εφαρμόζονται ε, σε περίπτωση ψηφοφοριών ε, βάσει των άρθρων 6 γάμα παράγραφος 2 7, ε, και 7 παράγραφος 3 6 και 8 σε περίπτωση ασυλίας βουλευτών. Σας ζητώ λοιπόν ζήτησε ο συνάδελφος κ. Μπρόντς το λόγο. Yes. Ναι. Κοιτάξτε, μια που μιλάμε για την άρση της ασυλίας, τα μέλη της Επιτροπής ε, θα ακούσουν μια συζήτηση και μετά θα ψηφίσουν. Στο σύνολο του Κοινοβουλίου το... η Ολομέλεια ψηφίζει αλλά δεν συζητά. Και έχουν εντύπωση πως το να γίνει ψηφοφορία χωρίς συζήτηση είναι στην καλύτερη περίπτωση κάτι το οποίο δεν έχει νόημα και στη ρότερη περίπτωση κάτι διαστραμμένο. Είτε δεν έχει δικαίωμα να ε, συμμετάσχει στην απόφαση του Κοινοβουλίου, οπότε δεν μπορεί να ψηφίσει ή αν ψηφίσει πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση για να ακουστούν τα επιχειρήματα. Αλλιώς μπαίνει κανείς στον πειρασμό να ψηφίσει με βάση προκαταλήψεις ε, αντί για πληροφορίες και στοιχεία. Ε, Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα με μια ερμηνεία και όχι αλλαγή του κανονισμού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως οι αποφάσεις ε, του Κοινοβουλίου σε ζητήματα ασυλίας ε, δεν είναι ουσιαστικές. Δηλαδή δεν κρίνουμε την αθωότητα ή την ενοχή του συναδέλφου. Απλά εγκρίνουμε στην Ολομέλεια την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής η οποία αφορά το παραδεκτό ή όχι της αίτησης ε, της αρμόδιας αρχής ε, του κράτους μέλους που έκανε το αίτημα και βεβαίως επιβεβαιώνουμε ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Οπότε οι αποφάσεις της Ολομέλειας είναι τεχνικές και απλές. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε σοβαρά για το αν θα παρεκκλίνουμε από το άρθρο του κανονισμού που λέει πως όλες οι τελικές ψηφοφορίες σε εκθέσεις στην Ολομέλεια είναι με ονομαστική ψηφοφορία. Αλλά οπωσδήποτε δέχομαι πως ε, για κάποιες ειδικά εθνικότητες ε, οι ψηφοφορίες για ζητήματα συλλίας είναι ευαίσθητες και πρέπει να το δούμε ρεαλιστικά το ζήτημα. Και άρα συμφωνώ με την διατύπωση που έχετε στην επιστολή σας ε, προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Αλλά επίσης θα πω πως ε, καθώς πλησιάζουμε στην επόμενη συνέλευση το όλο αυτό ζήτημα της κυριαρχίας του Κοινοβουλίου για ζητήματα προνομίων και ασυλίων ε, είναι κάτι που πρέπει να ξαναδούμε. Και βεβαίω η προηγούμενη μας απόφαση για το πρωτόκολλο του 1965 πρέπει να επανεξεταστεί. Και με ιδιαίτερη θέρμη θα έλεγα. Ωραία, λοιπόν, δεν βλέπω να ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Διανατασχερό ε, δεν χρειάζεται, πιστεύω. Δεν βλέπω να διαφωνεί κανένα. Ε, θα στείλουμε λοιπόν αυτή την επιστολή με το περιεχόμενο που μόλι σα διάβασα. Για το οποίο δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Ε, ψήφισαν υπέρ και οι συντονιστέ ομόφωνα. Τα αποφασίζουμε λοιπόν. Έχουμε τελειώσει και πρέπει να πω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Αυτά τα πέντε χρόνια εργασίας αυτήν την Επιτροπή ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Η Επιτροπή αυτή έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Δεν έχουμε πολλές νομοθετικές εξουσίες. Ωστόσο, τα καθήκοντά μας μας επιτρέπουν να συζητάμε χωρίς πολλές αντιπαραθέσεις με τρόπο επικοδομητικό και βάση λογικής. Είμαστε λοιπόν μια επιτροπή που κυριαρχείται από τις νομικές γνώσεις όλων μας και από μια βούληση να συνεργαστούμε. Εγώ εύχομαι σε όσους εξακολουθούν να είναι υποψήφοι για τις επόμενες εκλογές να επανέλθουν σε αυτά εδώ τα έδρανα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας. Να χαιρετήσω και τους νέους κράτες που βρίσκονται εδώ που μου δίνουν την ευκαιρία να μιλήσω για την Ευρώπη. Γιατί η Κροατία είναι η τελευταία χώρα που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η τελευταία χώρα, μια από τις τελευταίες χώρες που είχε μια αιματηρή εμπειρία πολέμου. Αν είχε μπει ίσως η Κροατία πρωτήτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχε υποφέρει από αυτή την καταστροφή. Η Ευρώπη γεννήθηκε για να αποτελεί μια ειρηνική ήπειρο και μια ειρηνευτική ήπειρο. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο. Εύχομαι λοιπόν σε αυτούς τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά σε, αυτή, την, σε αυτό το έργο το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θέλω να πει κάτι κύριος Ντάφ. Ευχαριστώ. Από πλευρά των συντονιστών στην Επιτροπή για αυτή, θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά για την προεδρία σας τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια. Πάντα ήσασταν ιδιαίτερα ευγενείς με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Ήσασταν γεμάτος ενθουσιασμό προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των εργασιών μας εδώ και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, κάτι το οποίο είναι πολύτιμο. Δεν συμφωνούσαμε πάντα μεταξύ μας, βέβαια, αλλά πάντα είχαμε διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και εσάς και το προσωπικό ειλικρινά για την εμπειρία αυτής της συνεργασίας που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ κύριο Σαπλή. Ευχαριστώ Είμαι αναπληρωτής, οπότε τι θα πω. Ευχαριστώ. Αλλά και εγώ ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την καρποφόρα πενταετία. Όντω είναι μια κάπως ιδιαίτερη η Επιτροπή μας. Καταφέραμε όμως να συνεργαστούμε καλά, να είμαστε πάντα φιλικοί μεταξύ μας. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ θετική εμπειρία. Η δουλειά γινόταν πάντα, μπορεί να μην συμφωνούσαμε πάντα μεταξύ μας, αλλά πιστεύω ότι και το δικό σας το έργο ήταν που βοήθησε πάρα πολύ. Γι' αυτό εκ μέρου όλων των μελών της Επιτροπής μας και αυτών που δεν είναι παρόντες εδώ σήμερα, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Ευχαριστώ. Όπως είπε ο κ. Νταφ, που γνωρίζει τα ευρωπαϊκά θέματα, θα πρέπει να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τη γραμματεία μας, διότι χωρίς τη συνεργασία της γραμματείας μας δεν θα μπορούσαμε να είχαμε εργαστεί τόσο σωστά, τόσο έγκαιρα και τόσο αποτελεσματικά. Τερματισμός της συνεδρίασης, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε με ποια έννοια, θα τα ξαναπούμε με έναν τρόπο διαφορετικό.